θα ε, συμφωνήσουμε. Θέλουμε να προχωρήσουμε, θέλουμε να βγουν οι ασυμμετρίες, αλλά είναι και το σύστημα πιο εύκολο. Ευχαριστώ πολύ.